Good afternoon to all of you, whether here... Καλησπέρα σε όλους σας, όσους βρίσκεστε στην αίθουσα και όσους μας παρακολουθείτε από την Ευρώπη, ακόμη και εκτός της Ευρώπης. Θα αναγγείλω τα αποτελέσματα της πρώτης χθεσινής ε, τροπολογίας, με ψηφοφορίες με τις τροπολογίες. Θα σας πω ποιες τροπολογίες έχουν γίνει αποδεκτές και ποιες απορρίφθηκαν. Οι τροπολογίες που δεν θα αναφέρω έχουν καταπέσει και όλοι έχετε λάβει τα συνολικά αποτελέσματα με τις ψήφους υπέρ, κατά και αποχές για κάθε ε, τροπολογία ξεχωριστά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες ε, για το τμήμα 3 του προϋπολογισμού 2020, ο εισηγητής είναι ο κύριος Λαρουτρού. Ε, πρώτο μπλοκ έχει ε, ε, εγκριθεί, το μπλοκ 2 έχει επίσης εγκριθεί το μπλοκ μείον 9 επίση έχει εγκριθεί. Τροπολογία 109 απορρίπτεται. Η τροπολογία 111 απορρίπτεται. Η τροπολογία 129 εγκρίνεται. Η τροπολογία 132 απορρίπτεται. Η τροπολογία 141 κατά τμήματα το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Η τροπολογία 145 κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα εγκρίθηκε. Η τροπολογία 147 εγκρίνεται. Η τροπολογία 150 εγκρίνεται επίσης. Η 182 εγκρίνεται. Η 209 εγκρίνεται. Η 210 εγκρίνεται. Η 220 εγκρίνεται. Η τροπολογία 229 απορρίπτεται. Η τροπολογία 234 απορρίπτεται. Η 245 εγκρίνεται. Η τροπολογία 246 εγκρίνεται. Το τρίτο μπλοκ εγκρίνεται. Η τροπολογία ΦΑΜ 6 εγκρίνεται. Η τροπολογία ΑΦΕΤ 17 εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στι τροπολογίε για το σχέδιο διορθωτικού Προπολογισμού 3 ε, του 2020 με εισηγήτρια την κυρία Μόνικα Χολμάγερ. Τροπολογία 1, 2 και 3 έχουν απορριφθεί. Περνάμε τώρα στις τροπολογίες για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού ε, Ταμείου Αλληλεγγύης για να παρασχεθεί ε, βοήθεια στην Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Αυστρία ο κύριο Φερνάνδε είναι ο εισηγητή. Τροπολογία 1 εγκρίνεται. Τροπολογία 2 εγκρίνεται. Περνάμε στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για προ... προηγούμενη έγκριση για το κτίριο Βάη στο Στρασβούργο. κυρία Κέλλερ ήταν εισηγήτρια. Εγκρίνεται το αίτημα για το κτίριο. Αυτά ως προς τις χθεσινές ψηφοφορίες και θα συνεχίσουμε με το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης, το τέταρτο σχέδιο, συνδευτικές προτάσεις για την παροχή βοήθειας στην Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και Αυστρία. Η κυρία Χολμάγερ είναι η συγγετριά για το σημείο 13 και της δίνω το λόγο για τρία λεπτά. Thank you very much. Can you hear me? Ευχαριστώ, με ακούτε. Σας ακούμε. Πολύ ωραία. Μιλάμε για το Ταμείο Αλληλεγγύης για το έτος 2020. Πορτογαλία καταρχάς. Με τον Τιφώνα Λορέντσο και τις Αζόρες ε, τον Οκτώβριο του 2019. Στη συνέχεια έχουμε την Ισπανία. Με πολλές πλημμύρες ε, Βαλένσια, Μούρσια, Καστιλιά, Αλαμάνκια και Ανταλουσία το Σεπτέμβριο του 2019, Ιταλία, Αυστρία, με ακραία καιρικά φαινόμενα και πολλαπλές πλημμύρες και άλλα ζητήματα με το έδαφος στην Ιταλία και εν μέρη στην Βενετία και στην Αυστρία στο Ανατολικό Τυρόλο. Το φθινόπωρο του 2019. Γι' αυτό λοιπόν προβλέπεται από την 13.06.01 να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Έχουμε εδώ λοιπόν, λοιπόν πληρωμές και δεσμεύσει σε ύψος 272 ε, εκατομμυρίων ευρώ. Θα προτείναμε λοιπόν να τα πρότεινα να υπερψηφιστούν αυτές οι προτάσεις. Ευχαριστούμε κυρία Χολμάιρ. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 14 της ημερήσιας ένταξη στο κινητοποίηση του EGF 2020 και να δώσω το λόγο στον κύριο Βίκτορ Νεκρέσκου, τον εισηγητή για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφε. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να βρούμε το σημαντικό έργο της Επιτροπής μας για το σημαντικό, τη σημαντική αρρωγή που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προς τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τον κορονοϊό. Και καταρχάς μιλάμε λοιπόν για την κινητοποίηση για του, του προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και τα δεύτερον να σας πω ότι όλοι ξέρουμε ότι το ΑΜΙΟ έχει ως σκοπό να δώσει αρρωγή σε εργαζόμενους και άτομα τα οποία υπέστησαν μεγάλες δυστατικές αλλαγές λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω της ε, συνέχισης ε, και εμβάθυνσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Να παράχθει, να παράχουμε λοιπόν ε, αρρωγή στους ε, ανθρώπους για να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Η έκθεση αυτή λοιπόν αφορά την κινητοποίηση εκατομμυρίων ευρώ από πλευρά ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα παρακολουθήσουμε την συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και θα παρέχουμε αρρωγή στα κράτη-μέλη για την υλοποίηση του Ταμείου. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε κάποια βασικά σημεία του Ταμείου σε ό,τι αφορά την ορατότητα, την προβολή του προγραμματός σε όλα τα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά και την, ε, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη τη διαδικασία, αλλά και να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Πέραν αυτών, συμφωνήσαμε και σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους μας ε, από την Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί διευκρινίσαμε κάποια σημαντικά στοιχεία. Και αυτά πλέον καταγράφονται στην έκθεση ότι σύμφωνα με τους τρέχοντες κανένους το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους αυτοαπασχολούμενους στο πλαίσιο της ε, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από το COVID-19. Και αυτό είναι σημαντικό λοιπόν ότι αναφέρεται πλέον στο φάκελο αυτό με την υποστήριξη τη Επιτροπή και τη Γραμματεία. Σα ευχαριστώ λοιπόν συναδελφοί για την δουλειά σα και ελπίζουμε να υπάρξει ευρεία πλειοψηφία υπέρ τη πρόταση, αλλά και μεγάλη συμμετοχή προκειμένου να πετύχουμε πραγματικά την ευρωπαϊκή ανάκαμψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκρέσκου. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 15 για το τμήμα 2 των μεταφορών ή το 2020 και να δώσω το λόγο στην συγγήτρια την κυρία Χόλμαϊερ. So, ich hoffe, ihr könnt mich wieder hören. Herzliche Grüße noch. Ελπίζω να με ακούτε. Χαιρετισμούς από την Βαβαρία. Έχουμε το D4 τεχνική αρρωγή σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μιλάμε για 345.000 ευρώ. Μετά έχουμε το ΤΕΚ 9. 15,8 εκατομμύρια ευρώ από την ε, γραμμή 32030202 γρήγορα και αποτελεσματικά μέτρα σε καταστροφές μεγάλης κλίμακας σε τρίτες χώρες στη γραμμή 230201 για διάθεση ε, γρήγορης ανθρωπιστικής βοήθειας και επισητιστικής βοήθειας. Η Κομισιόν ήδη είχε διαθέσει το ποσό αυτό στο μηχανισμό βοήθειας ε, καταστροφών γιατί ήταν απολύτως ε, ανάγκη να έχουμε την αλλαγή του προϋπολογισμού 21-2020 η οποία εγκρίθηκε στις 17 Απριλίου του 2020 και η Κομισιόν ζήτησε την χρήση αυτού του μέσου για σκοπούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Το τελευταίο σημείο αφορά την μεταφορά DEC 10 η οποία αφορά 55,9 εκατομμύρια ευρώ στην γραμμή 230201 για την άμεση παροχή ανθρωπιστικής και επιστημιστική βοήθειας από την γραμμή του προϋπολογισμού βελτίωσης 190401 ε, και από την αναπτυξιακή βοήθεια τη γραμμή για τη συνεργασία με την Ασία 27,9 εκατομμύρια, τη Μέση Ανατολή 10 εκατομμύρια και το Αφγανιστάν 15 εκατομμύρια. Τα κονδύλια θα διατεθούν στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας για τον COVID στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη, αλλά και στο Πακιστάν, Ιράκ και Αφγανιστάν. Όλες αυτές οι μεταφορές είναι εντάξει. Ε, προτείνω να υπερψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο σημείο 16 της ημερησίας διάταξης, μεταφορές του 2020 άλλα τμήματα. Πριν δώσω τον λόγο στην κυρία Γκουαρτία Θάμπαλ, να επισημάνω πως και οι οδησηγητές έχουν ήδη λάβει απαντήσεις ε, μέσω email σε κάποια από τα γραπτά ερωτήματα που απευθύνθηκαν προς τις υπηρεσίες ε, του Κοινοβουλίου τις προηγούμενες μέρες. Κυρία Γκουαρτία Θάμπαλ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε- οι σκιώδεις ηγητές έχουν ήδη τις απαντήσεις, οπότε δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Δύο μεταφορές έχουμε. Πρώτη είναι η C1 για το Κοινοβούλιο, 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια για να... Για την... Ε, Και για τις ε, συμπληρωματικές επενδύσεις σε τεχνολογία και πληροφορική που οπωσδήποτε χρειαζόμαστε με τα νέα δεδομένα της κρίσης COVID-19. Και οι μεταφορές για τις γραμμές αυτές προέρχονται από τα ταξιδιωτικά, συνήθι ταξιδιωτικά έξοδα για τις αποστολές που έχουν μείνει αχρησιμοποιητά, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τις τηλεδιασκέψεις. Η δεύτερη η C2 μεταφορά αφορά 1.800.000, ε, πάλι αφορά εργασίες ε, σε σχέση με το σύστημα πληροφορίας, τεχνολογίας της πληροφορίας και πρόκειται για μια επέκταση του ισχύοντος ε, συστήματος διαχείρισης χρηματοοικονομικής που υπήρχαν στο στον προπολογισμό και θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη κατανομή. Αυτές είναι οι δύο μεταφορές, η 1 και η 2, 11 εκατομμύρια και ένα 800 αλλά όπως είπα οι σκιώδεις ηγητές έχουν ήδη λάβει όλες τις απαντήσεις από τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω την ευγενική σας πρόσκληση. Αν υπάρχουν συμπληρωματικές ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, τώρα είναι η ώρα για να υποβληθούν. Κανένας ούτε εντός ούτε εκτός της δεν ζήτησε το λόγο, οπότε μπορούμε να περάσουμε στην έναρξη της δεύτερης ψηφοφορίας. Καταρχήν να ελέγξουμε αν συγκεντρώνουμε την απαρτία των 11 μελών, που είναι απαραίτητη για την έγκυρη ψηφοφορία. Παρακαλώ, πατήστε όλοι το κουμπί Raise Hand για να εξακριβώσουμε αν έχουμε την απαρτία. Στην πλατφόρμα Interaction πατήστε το κουμπί Raise Hand. It seems that we are uh, largely... Φαίνεται ότι έχουμε υπερβεί κατά πολύ τις απαραίτητους 11 σε συναδέλφους που είναι απαραίτητοι για την απαρτία. Έχουμε απαρτία υπέρ των δεών λοιπόν. Και από τη στιγμή που έχουμε εξακριβώσει την απαρτία να περάσουμε στη δεύτερη σύνοδο ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε τις τελικές ψηφοφορίες τη έκθεση για τι κατευθυντήριε γραμμέ για το τμήμα 3 του προπολογισμού του 2021. Επίση, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 3 κινητοποίηση του ΕΣΕΦ για την παροχή βοήθεια στην Πορτογαλία, Αυστρία, Ισπανία και Ιταλία, το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 4 και την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Επιπλέον, θα έχουμε και ξεχωριστές ψηφοφορίες για τα ακόλουθα θέματα. Καταρχήν, το ΔΕΚ 04 22 09 και επίσης το C, τις μεταφορές C1 του 2020 και C2 του 2020. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 5 παρατέταρτο και θα διαρκέσει μέχρι τις 6. Έναρξη της περίοδου ψηφοφορίας σημαίνει σε αυτούς τους καιρούς που διαβιούμε και κήρυξη του τέλους της συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε αργότερα.